12.30. Θα πρέπει να σας διαβάσω μια ανακοίνωση. Οι φιλανδικές αρχές κοινοποίησαν ότι ο κύριος Πεντήλα ορίστηκε ευρωβουλευτής αντικαθιστώντας τον κύριο Ιτάλα από την 1η Μαρτίου 2012. Κατά συνέπεια, ο κύριος Πεντήλα Τίλα παρετήθηκε από Ευρωβουλευτής από την 1η ε, Τρίτου 2012. Σύμφωνα με τον κανονισμό, το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη ότι η θέση χειρεύει από την ημερομηνία εκείνη και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.